Ladies Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Ε, υιοθέτηση της ημερησίας διατάξεως. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη, οπότε εγκρίνεται. Νομίζω ότι θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το διευρυμένο Προεδρείο θα συνεδριάσει ε, στο τέλος συνεδριάσεως μετά με, από την ανταλλαγή απόψεων με τον James Morrow σχετικά με την κατάσταση στο Κάιρο. Έχουμε λες επίσης τον κύριο Λιάν και Υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας για να έρθει στις 31 Μαρτίου αν συμφωνείτε και στις 21 Μαρτίου θα θέλαμε να κάνουμε μία συζήτηση σχετικά με την ε, ε, ίδρυση της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η την περασμένη εβδομάδα είχα συζήτηση με τον κύριο Κόπλερ εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Ιράκ και μας ενημέρωσε για την κατάσταση στο Ιράκ και επίσης για την ε, κατάσταση στο Καμπ Ασάφ εάν, στο στρατόπεδο ΑΣΑΦ. Οπότε εάν συμφωνείτε θα ε, ε, σας ενημερώσω για αυτό το θέμα διότι ε, είναι ένα θέμα που χειρίζεται ο εκπρόσωπος του ο Αμερικανού Προέδρου και η κυρία και η νέα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Ιράκ επίσης θα έπρεπε να έρθει αν μπορεί. Ερχόμαστε στο τρίτο θέμα, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση πρόοδου για τη Βοσνία Εζεργοβίνη 2011. Ε, η ομιλήτρια είναι η κυρία Ντόρι Σφάκ, είναι η συγγήτρια. Έχουμε καθορίσει και συμφωνήσει ότι η προθεσμία τροπολογιών είναι 9 Φεβρουαρίου στις 12 και αν συμφωνούν οι συνάδελφοι θα παραμείνουμε με αυτή την ημερομηνία και η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, είναι αξιοπερίεργο ότι σχετικά με την έκθεση πρόοδου για το προηγούμενο έτος μόνο τώρα ε, γίνεται η παρουσίαση γιατί μέχρι το Δεκέμβριο δεν έγινε τίποτα καινούριο, δεν είχαμε κυβέρνηση, η κατάσταση είχε σκληρίνει και λίγο πριν το τέλος του χρόνου διαπιστώσαμε ότι οι πολιτικές, τα κόμματα μπόρεσαν να καταρτήσουν μια κυβέρνηση η οποία όμως ακόμη δεν έχει συσταθεί και ε, πρόεδρος θα είναι ε, ο κύριος Μπεβάντερ τίποτα άλλο όμως δεν είναι σαφές αλλά οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων συμφώνησαν επί ορισμένων πολιτικών θεμάτων και εν Σχέση με ό,τι έχω στην έκθεσή μου που λέω ότι από την Παρασκευή υπάρχει και ε, ένας νόμος για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να σας πω ε, ότι θα πρέπει να τροποποιήσω προς το θετικό την έκθεσή μου πριν ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Διήρκεσε όμως πολύ και ακόμη διαρκή μέχρι ότου να, μπορέσω, ε, να μπορέσει να συσταθεί μια κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα διότι δεν υπάρχουν επαρκείς ε, συμβιβασμοί και συνενητική πρόθεση εις ε, την ε, υπερισχύουσα πολιτική παράταξη και δεν υπάρχει θέληση να καταλήξουν κάπου. Οπότε είδαμε ότι πέρυσι ναι μεν δόθηκε ελευθερία θεωρήσεων κατόπιν όλης της πιέσεως οι οποίες υπήρχαν και οι κυβερνώντες αντελήφθησαν ότι δεν μπορούσαν παρά να συνεργαστούν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρόμαστε που μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη Έχουμε επιτέλους έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αρχηγό της αντιπροσωπείας και πέραν από αρχηγός της αντιπροσωπείας είναι ο ε, ε, εντεταλμένος ε, ο εκπρόσωπός μας σαν πρέσβη στην περιοχή την οποία γνωρίζει από ετών πολύ καλά και προσπαθεί ε, επί τόπου να συνεννοηθεί με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με τα πολιτικά κόμματα και να ξεκινήσει μια θετική διαδικασία. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι ότι το κράτος έχει ε, διαρθρωθεί σε δύο οντότητες οι οποίες αποτελούν αποτελούν το συνολικό κράτος. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς είναι δυνατόν και στις δύο οντότητες αυτές να μην υπάρχει κατανόηση για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο κράτο και δεν μπορεί ε, κάθε οντότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα. Όσο οι οντότητες νομίζουν ότι κάτι θα χάσουν, ότι η οντότητά τους θα τους υφαρπαγεί εάν ε, ε, προωθήσουν ένα σύγχρονο κράτο θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα διότι ορισμένα πράγματα μπορούν να διαπραγματευτούν μόνο ε, διακρατικά και η Βοσνία Ριτσεγοβίνη μπορεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εάν ε, υπάρχει μία διοίκηση η οποία λειτουργεί εν ονόματι ε, ολοκλήρου του κράτους και μπορεί να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πολλά προβλήματα. Καταρχήν τη διαφθορά που είναι σαν ένα καρκίνωμα στην περιοχή και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ε, πολύ αποτελεσματικά και ε, ε, πρέπει να πούμε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη όσον αφορά τα, τα εγκλήματα πολέμου συνεργάζεται με το Διεθνές Δικαστήριο αλλά όσον αφορά την παρακολούθηση και την δίωξη των εγκληματιών πολέμου πολέμου επιτόπου χρειάζεται να γίνουν προόδοι και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι ο ε, νομικός και δικαστικός μηχανισμός δεν λειτουργεί στη Βοσνία Ζεγοβίνη παρόλο που πιέζουμε εδώ και χρόνια ασχολήθηκε ακόμη και η Λέιντι Άστον και ε, ε, διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Ρεπούμπλικα Σέρψα θα υπάρξει ένας σωστός διάλογος ε, δεν, ε, η ε, Ρεπούμπλικα Σέρσφα δεν δέχεται αυτή τη δικαιοσύνη αλλά χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να αναγνωριστεί ένα κράτος. Άρα αυτό το οποίο επιζητείτε με αυτό το διάλογο είναι θετικό αλλά πρέπει κάπου να καταλήξει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε πάντοτε όταν υπάρχει μία δικαστική μεταρρύθμιση είναι ότι οι εγκληματίες πολέμου για ό,τι διαδραματίστηκε στη Βοσνία Ερδεγοβίνη δεν έχουν τύχει σωστή αντιμετώπιση και τα θύματα μέχρι σήμερα δεν έχουν, δεν μπορούν να πούμε αποζημιωθεί αλλά δεν ξαναβρήκαν το δίκιο τους. Οπότε ο ένας ε, ε, μετακυλεί στον άλλο τις ευθύνες ε, και εδώ πρόκειται ως επτοπλίστων για γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές λοιπόν πρέπει να βρουν το δίκιο τους κάποτε η συνεχής επιστροφή, η εσωτερική διακίνηση είναι κάτι το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί και εγώ πιστεύω ότι αν έχει κανείς προσυπογράψει τη διακήρυξη του Σιράγεβο για τους πρόσφυγες πρέπει να τη σεβαστεί και γι' αυτό με τους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο της Βοσνίας το έχουμε συζητήσει διότι η διακήρυξη του Σαραγεύου είναι σημαντική και όσοι πρόσφυγες θέλουν να επιστρέψουν πρέπει να μπορούν να το πράξουν. Θέλω να σας πω αυτό το οποίο δεν ξανάγραψα στην έκθεση το οποίο όμως έχω γράψει σε όλες μου τις εκθέσεις ότι στο βορρά στην, περίοδο, στην περιοχή Ποσαβίνα η εικόνα είναι ίδια όπως αμέσως μετά τον πόλεμο τίποτα δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει επικοδομητικά κανείς δεν επιστρέφει και όσοι επιστρέφει Όποιος επιστρέφει και χτίζει ένα σπίτι δεν μπορεί να έχει ούτε ηλεκτροδότηση ούτε νερό οπότε μπορούν να κλείσουν το σπίτι και να ξαναφύγουν παρακαλώ το, την Ρεπούμπλικα Σέρψα να κάνει κάτι και μου λένε μα εγώ είμαι μόνο πρόεδρος πρέπει να ρωτήσουμε τις κοινότητες θα έπρεπε όμως οι άνθρωποι να μπορούν να επιστρέψουν εκεί που θέλουν στο θέμα της εκπαιδεύσεως μπορούν να γίνουν ακόμη πολλά. Είναι πολύ δυσάρεστη κατάσταση, ιδίως για αυτούς που εργάζονται ε, ε, τους, στο θέμα της παιδείας. Είχαμε 13 υπουργούς ε, εκπαιδεύσεως, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Βοσνία ζεγοβαίνει σε σχέση με το 2007 δηλαδή αυτά που προσφέραμε το 2007 δεν μπορεί να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους νέους γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να δημιουργήσουν έναν οργανισμό που θα το διαχειριστεί. Οπότε δέστε τη Βοσνία όπου υπάρχει ελάχιστη ελπίδα για τους νέους σας υπενθυμίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μία εσωτερική αγορά η οποία καλώς ή κακώς λειτουργεί. Ε, δεν υπάρχει όμως καμία εσωτερική αγορά μεταξύ Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Εάν τα σύνορα αυτά δεν καταργηθούν τότε και η χώρα δεν θα μπορέσει να προοδεύσει. Πρέπει λοιπόν αυτά να γίνουν επιτόπου για να υπάρξει προκοπή. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ε, θυμάστε την ε, πτώση Φίντσι ε, η οποία υπάρχει εις τη συνθήκη του Ντέιτον όπου υπάρχουν ε, τρεις ε, εθνότητες εκ των οποίων η μία δεν μπορεί να συμμετάσχει εις τις πολιτικές διαδικασίες ή υπάρχουν και άλλοι Ρωμά και άλλες εθνότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται σαν άλλη, διαφορετική. Και ε, το δικαστήριο αποφάσισε στην περίπτωση Φίντσι ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Εις ε, το κοινοβούλιο των Ρώμα ε, υπήρξε μία διαβούλευση και προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα χωρίς να επέμβει η διεθνής κοινότης, πράγμα το οποίο εύχομαι μακάρι να μπορέσουν να κάνουν κάνουν τις δουλειές τους και να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις τους μόνοι τους και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προσπαθεί να κάνει ομάδες εργασίες και να τις αφήσει να εργαστούν επί του θέματος μόνες της τι άλλα προβλήματα όμως έχουμε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πάρα πολλά. Ανέφερα μερικά. Αλλά θέλω να επανέλθω στην ε, ε, εκπαίδευση διότι η κατάσταση υπάρχει και σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου δημιουργούνται ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία ζητούν πολλά χρήματα για τις σπουδές, το περιεχόμενο περιεχόμενο της διδασκαλίας είναι ελάχιστο και το τέλος δεν μπορεί κανείς να αξιοποιήσει αυτά τα διπλώματα. Υπάρχουν accreditation agencies, δηλαδή οργανισμοί διαπιστεύσεως και πιστοποιήσεως και αντί να δίνουμε τα χρήματά μας για διπλώματα που δεν θα οδηγήσουν πουθενά, εάν συνεργαστούμε με το νομικό τμήμα της Μπάνια Λούκα πρέπει να σας πω ότι αν το συγκρίνουμε με μία ε, άλλη χώρα η ποιότητά του είναι πάρα πολύ χαμηλή και πρέπει να βελτιωθεί. Ένα άλλο θέμα είναι ότι στη χώρα αυτή δυστυχώς ο ΩΣΑ ε, είχε δημιουργήσει δύο σχολές από κοινού όπου από τη μία πλευρά ε, ε, φοιτούν οι μουσουλμάνοι και από την άλλη μεριά οι Κροάτες πράγμα το οποίο είναι μεσαιωνικό τα παιδιά τα οποία συνηθίζουν από μικριά ε, ότι είναι διαφορετικά δεν μπορούν να διαιωνίζονται σε μια τέτοια κατάσταση διότι η συνειδητοποίηση αυτή ξεκινά την πρώτη χρονιά που πάνε σχολείο και θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να καταργήσουμε αυτές τις ε, χολές και να τις συγχωνεύσουμε σε μια ενιαία τάξη όπου τα παιδιά θα φοιτούν μαζί. Ε, επίσης η διοίκηση είναι τραγική. Όχι μόνο υπάρχει ε, τεράστια διαφθορά αλλά υπάρχει και τεράστια ε, διοίκηση. Σας μίλησα για 13 Υπουργεία παιδείας για να καταλάβετε. Θα τα αναφέρω αυτά στην έκθεσή μου, αλλά ουσιαστικά είπα ότι ε, όλοι το γνωρίζουν ότι το έχω διακηρύξει και δεν με συμπαθούν, αλλά η Ομοσπονδία αυτή έτσι όπως έχει καταρτιστεί ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχει 10 καντόνια, έχει την τοπική αυτοδιοίκηση, μετά 10 φορές 10 υπουργούς, την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, κυβέρνηση και μετά ε, πάνω από αυτήν την κρατική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Καταρχήν υπάρχουν 140-150 υπουργοί. Δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά ακολουθούν μία κατεύθυνση η οποία δεν έπρεπε να ακολουθείτε. Πρέπει να επενδύσουμε στη νεολαία και σε κοινωνικές δομές και όχι σε θεσμούς οι οποίοι εμποδίζουν ο ένας να λειτουργήσει ο άλλος. Τα προανέφερα όλα αυτά και ε, κάτι πρέπει να γίνει πολλοί μου λέγουν πώς αντιμετωπίζετε τον ύπατο εκπρόσωπο. Ο πρώτος ύπατος εκπρόσωπος ήταν ο κύριος Μπίλντ. Η γυναίκα του ήταν συνάδελφος και τώρα είναι υπουργό εξωτερικών της Σουηδίας. Ήταν ο, ο κύριος Μπίλντ ο πρώτος ο οποίος μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε ε, και το έπραξε ε, προσπάθησε προσπάθησαν να υπάρξει ένα, μία, ένα ενιαίο διαβατήριο που δεν είχαν πετύχει οι ντόπιοι πολιτικοί, να υπάρχει εθνικό σήμο, σημαία, ε, τα σύμβολα του κράτους και έχει νομοθετήσει πολλά διατάγματα. Αλλά σήμερα είμαστε σε μία κατάσταση όπου ο, εκπρόσωπος, ο, ο ύπατος εκπρόσωπος αυτός δεν θα έπρεπε πλέον να παραμένει διότι με την παρουσία σου του και μόνο επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένας τέτοιος θεσμός ο οποίος δεν είναι αποδεκτός σε ένα κυρίαρχο κράτος ότι ένα τέτοιο θεσμός εμποδίζει τους πολιτικούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος αποφασίζει, γιατί τότε εγώ να αποφασίσω και να ε, θυμώσω τους ψηφοφόρους μου. Γι' αυτό και είπα ότι θα έπρεπε να δούμε εάν αυτός ο ύπατος ε, εκπρόσωπος δεν αποσυρθεί σιγά σιγά. Ολισμένοι έχουν αντίθετη άποψη, αλλά εγώ ε, είμαι υπέρ ε, του, της πιο αυστηρής αντιμετώπισης. Πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν, πολλά έχουν ήδη δρομολογηθεί. Και αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι υπάρχει ένα τρίτο μέρος εκτός από τις δύο οντότητες αυτές στον Βορρά υπάρχει η περιοχή Μπρίτσφο όπου και οι τρεις επεμβαίνουν που είναι κάπως κατοχυρωμένο και το οποίο έχει μία δομή την οποία όλοι στηρίζουν. Όσον αφορά τη διμερή συνεργασία στην περιοχή δεν πάμε κακά η Βοσνία Ζεγοβίνη δεν έχει άμεσα προβλήματα με τις ε, τα γειτονικά κράτη ε, υπάρχει μία συνεργασία που επιλύεται ε, με την Κροατία για την περιοχή ε, γύρω από τον Ντουμπρόβνικ διότι ένα κομμάτι της Κροατίας μπαίνει μέσα στην άλλη χώρα δεν ξέρω για πόσα χιλιόμετρα είναι 10 χιλιόμετρα που περνά κανείς από τη Βοσνία για να επανέλθει στην Κροατία χρειάζεται μία γέφυρα υπάρχουν συζητήσεις αλλά με καλό πνεύμα θα μπορέσει το πρόβλημα να επιληθεί μεταξύ των δύο χωρών. Και η Κροατία σαν άμεσος γείτονα το 2013, στο μέσο του 2013 θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και για τη Βοσνία θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα διότι θα υπάρχουν ε, σύνορα που δεν θα μπορεί να υπερβεί ιδίω στον τομέα που θα έπρεπε να μπορεί μπορεί να τα επιλύσει όσον αφορά τα τρόφιμα, τα γεωργικά προϊόντα και εδώ και 10 χρόνια παρακαλούν γονατιστή, ε, παρακαλούμε γονατιστή να ψηφίσουν τη νομοθεσία για τα υγειονομικά θέματα και ε, εάν αυτό δεν γίνει θα έχουν οι επιχειρήσεις της Βοσνίας Ευζεγοβίνης σοβαρά προβλήματα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον όσον αφορά την διατροφική ασφάλεια θα μπορέσουμε να έχουμε μία πρόοδο που θα είναι και προς του κράτους. Όλα αυτά λιγάκι άτακτα σας τα παρουσίασα. Μπορείτε όλοι να διαβάσετε την έκθεση και στη συνέχεια να διατυπώσετε ιδίαν γνώμη. Και ο πρόεδρος νομίζω ότι θα διαβάσει την έκθεση, οπότε εφόσον έχω το κείμενο γερμανικά δεν χρειάζεται ο κύριος Μπρόκ μιλάει συνέχεια αγγλικά. Οπότε όλοι οι συνάδελφοι θα διατυπώσουν ιδία γνώμη και στη συνέχεια μπορεί σε ένα ή δύο σημεία να βελτιωθεί, να γίνει πιο εχμηρό το κείμενο, αλλά εάν το αποδυναμώσουμε δεν θα μας ακούσουν. Με τη διπλωματική γλώσσα, τη φλιαρία δεν θα προχωρήσουμε, δεν μας ακούνε, δεν μας πιστεύουν και πιστεύω ότι σαν κοινοβούλιο πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν είμαστε εμείς διδάσκαλοι, ε, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει μαζί με τους πολιτικούς να επέμβει σε αυτές τις περιοχές για να μην μείνει η πολιτική κατάσταση ένα βήμα πριν από την κατάληξη. Όλα αυτά θα έπρεπε να διορθωθούν, αλλά χρειάζεται και προθυμία των πολιτικών κάτι να κάνουν πράγμα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο μέχρι τώρα αλλά νομίζω ότι το νέο έτος ξεκίνησε καλύτερα από ό,τι τέλειωσε το προηγούμενο. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Κοιτάξτε, ε, υπάρχει ένα θέμα, σε ένα θέμα όπου υπάρχει μια χώρα που είναι χειρότερη από την Βοσνία Σεχοβίνη όσον αφορά τουλάχιστον τον αριθμό των Υπουργών Παιδείας. Αναφέρομαι στη χώρα μου. Στη Γερμανία έχουμε 17 Υπουργού Παιδείας και εκεί τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Η κυρία Πακ, ναι, αλλά όχι 17 υπουργού ε, στη Βόρεια Ερναβία εκεί έχουμε μόνο ένα. Και αυτός περισσεύει, λέει ο πρόεδρος, χαριτολογώντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την έκθεση αυτή ε, που είναι μια έκθεση νυφάλια Ελπίζω λοιπόν ότι επιτέλους ελπίζω να γίνει κάτι. Αλλά βεβαίως ε, πρέπει να υπάρχει και επιθυμία για, βοήθεια, για αυτοβοήθεια. Να θέλουν και εκείνοι να δεχθούν τη βοήθεια και να βοηθηθούν μόνοι τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην κυρία Πακ, διότι είναι πάρα πολύ αξιολογική η και επίσης την ευχαριστούμε διότι μας έδωσε μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη εισαγωγή Όσον αφορά τώρα την έκθεση, φύγει όλα τα σημαντικά θέματα. Επίσης, είναι πάρα πολύ εύστοχη η γενική έποψη της καταστάσεως την οποία μας έδωσε και συμφωνώ με την εισηγήτρια προσωπικά ότι δυστυχώς είχαμε μόνο πολύ συγκεκριμένη, περιορισμένη πρόοδο στα περισσότερα των ε, σημείων που αφορούν την υπόθεση αυτή και γι' αυτό και είναι ουραγός σχέση με τις υπόλοιπες ε, χώρες της περιοχής η Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί εδώ, όμως η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη όσον αφορά αυτό το πρόβλημα. <clears throat> και κοιτάξτε, πρέπει επιγόντως η χώρα να επιδείξει μια ικανότητα ευρωπαϊκής προσαρμογής, το οποίο δεν θα καταστεί αυτό παρά μόνο αν δεν έχουμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, τους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα της ε, διοίκησης και ε, έχουμε μια γενική συμφωνία όλων των εμπλεκομένων ε, και αυτό ίσως θα ήταν ένα σημάδι ότι τα πράγματα μπορούν να σημειώσουν μια πρόοδο στη χώρα. Επίσης σημειώνεται μια πρόοδο όσον αφορά την εναρμόνιση του συντάγματος με ε, την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστή της Επιτροπής μάλλον των, Ευρωπαϊκών, των δικαιω, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα θα πρέπει να συμμεθούν ε, προσπάθειες και πρόοδος ε, στην δικαιοσύνη συγκεκριμένα, να υπάρξει κράτος δικαίου περισσότερο, να υλοποιηθεί μια διοικητική μεταρρύθμιση το οποίο δεν θα είναι δυνατόν παρά μόνο εάν το αναλάβουν ως δική τους προσωπική ευθύνη οι Βόσνοι πολιτικοί και οι οποίοι θα πρέπει να αγκαλιάσουν, να ενστερνιστούν αυτή τη διαδικασία του εξευρωπαϊσμού, ούτω ώστε να μπορέσουν να λάβουν τι ευθύνε του για το μέλλον τη χώρα. Επίση, έχουμε το θέμα τη διεθνού εποπτεία επί τη χώρα, διότι συμφωνώ ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να πασχίσουμε προ εξέβρεση λύση, ούτω ώστε να υπάρξει περισσότερη ευθύνη, περισσότερη ανάληψη ευθύνη όσον αφορά την λειτουργία τη χώρα. Έχουμε και άλλα θέματα ε, επίγοντα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, τώρα στην ε, αμέσως επόμενη περίοδο και επίσης ε, εγώ ελπίζω ότι με τη νέα κυβέρνηση θα σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων και αυτό δεν είναι θέμα μόνο του, του, του πώς θα πλησιάσει την Ευρώπη η χώρα. Αυτό θα ωφελήσει πρώτα-πρώτα τον ίδιο το λαό της χώρας. Και σας ευχαριστώ.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 Eh, we zitten natuurlijk in een periode na een lange impasse wat betreft Bosnië en Herzegovina. Είναι αλήθεια, ε, χωρί να χρειάζεται να σα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η συγκήτρια, εγώ από σοσιαλιστών πρέπει να σα πω ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, μετά από αυτή την μακρά περίοδο ε, που πέρασε, τώρα βλέπουμε να υπάρχει μετά την αδράνεια μια μικρή πρόοδο. Οπότε και βλέπουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα αρχίσει να πράττει τα αναγκαία. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα ένα ένα αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο και επίση βλέπουμε ότι υπάρχει συμφωνία όσον αφορά, όπως προαναφέρθηκε, τον καινούριο νόμο περί της απογραφής και στατιστικής. Δηλαδή δεν πρέπει να προσέξουμε και ιδιαίτερο στο κεφάλαιο 7 όσον αφορά την επιστροφή των εκτοπισμένων. Είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό και θα αποτελέσει και κριτήριο για την πρόοδο. Επίση θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την αναθεώρηση του συντάγματο, Το έχει αναλάβει το κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή, θα πρέπει να δούμε τι τροπολογίε θα κατεβάσουν. Τέλος πάντων θα τα εξετάσουν αυτά. Επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι είπε το Συνταγματικό Δικαστήριο όσον αφορά τα προβλήματα συμβατότητας, όσον αφορά τα θέματα διπλής ηθαγένειας των υπηκών της χώρας, αλλά και όσον αφορά τους εκτοπισμένους. Δεν πέρασε το σχετικό νομοσχέδιο, αλλά θα πρέπει τελικά να επιλύσουν το πρόβλημα. Επίσης πρέπει να δούμε και τι έγινε με τα θύματα των σεξουαλικών εγκλημάτων ε, κατά τον εμφύλιο. Πριν από περίπου ένα-ενάμιση χρόνο, εγώ, η κυρία Σκούκα και η κυρία Πακ ε, απευθύνουμε μια επιστολή στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και στην κυβέρνηση της χώρας και νομίζω ότι πετύχαμε κάποια πράγματα, διότι μετά την επιστολή μας υιοθετήθηκε μια νέα στρατηγική. Να γίνει κάτι επιτέλους για αυτά τα θύματα. Μιλάμε για πάνω από 10.000 γυναικών που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Άρα το πρόβλημα είναι υπαρκτό και τελικά θα πρέπει να υιοθετηθεί κάποια κριτική. Ε, ε, βέβαια θα πρέπει να πιστούν και οι Σέρβο-Βόσνοι να προσχωρήσουν σε αυτές τις προσπάθειες. Αυτό βέβαια και εντάσσεται στο ζήτημα της προσέγγισης και της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013 η Κροατία θα καταστεί κράτος μέλος. Έχουν πολλά, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρων κοινών συνόρων οι χώρες και οπότε θα αναγύψουν ζητήματα εμπορικά και άλλα για τα οποία θα πρέπει το συντομότερο να επιτευχθεί συμφωνία. Προς το παρόν αυτά θέλω να σας αναφέρω όσον αφορά τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Περιμένουμε πώς και πώς τη συνέχεια της ε, θετικής μας εργασίας με την κυρία Πακ Κορνέλισεν. Η κυρία Κορνέλισεν, ευχαριστώ. Γενικώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αρκετά αξιόλογη αυτή η έκθεση και είναι πάρα πολύ θετικό ότι μπόρεσε η κυρία Πακ να διαπιστώσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Μας εξήγησε πού έχει σημειωθεί αυτή η πρόοδος, ενθαρρυντικά όλα αυτά και ενθαρρυντικό ότι ε, έχουμε γεγονός πέρασε το νομοσχέδιο για τις κρατικές ενισχύσεις. περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με στατιστική και ε, απογραφή αλλά θα πρέπει να δούμε πώς στην έκθεση θα εξισορροπήσουμε ότι από την άλλη μια μια αργία να μην είμαστε αισιόδοξοι ούτε όμως και αφελείς και από την άλλη να μην είμαστε καταστροφολόγοι και άκρος αρνητικοί. Ιδίω με ανησυχεί η κατάσταση σε σχέση με την δικαιοσύνη. Αυτό έχει καταστεί μέσω εκβιασμού, όπως είπαμε υπονομεύονται οι θεσμοί, το στεγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει δηλαδή και τόσο πολύ κράτο δικαίου και άρα θα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή αυτής της ε, υπονόμευσης των παραδοσιακών θεσμών και θεσμικών οργανών της χώρας. Θα πρέπει επομένω ο δομημένο διάλογο με τη χώρα να αποδώσει καρπού. Δεν ξέρω αν ο κ. Σόρτζεν ε, είναι στο πλευρό μας θα πρέπει το, η προνταξιακή διαδικασία να πλαισιωθεί με εντονότερη παρουσία μας σε διάφορες περιοχές της χώρας, ούτως ώστε να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο είδους αναβάθμιση θεσμική, αλλά και της δικαιοσύνης. Θα πρέπει και εμείς και άλλοι διεθνείς φορείς να έχουμε ενιαίο μέτωπο. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Η στάση της Ένωσης δεν διακρίνεται από ενιαία φωνή. Δεν έχουμε συνέπεια στην πολιτική μας. Οι εκπρόσωποι μας εκεί δεν συνειδητοποιούν το ρόλο του Σόρενζεν. Επομένως, πρέπει να σας πω ότι θα κατεβάσουμε κάποιες τροπολογίες σε σχέση με αυτά τα οποία σας εξήγησα και όπου θα διατυπώνουμε τις ανησυχίες μας. Γιατί με ευχολόγια η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί στη Βοσνία. Και ελπίζουμε ότι είναι επικοδομητική η κριτική που ασκούμε όσον αφορά τον διαρθρωμένο δεδομένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα και ότι η νέα κυβέρνηση θα δώσει κάποια όθηση ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος Πούζεκ έχει λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, όπως το έπραξαν και άλλοι. Νομίζω ότι η εκτεσή της είναι πολύ καλή. Ε, η εισηγήτρια αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στην ενθάρρυνση αφενός και αφετέρου στην αναγκαιότητα να εκπληρωθούν υποχρώσεις γιατί υπάρχουν, έχουν ήδη αναλυθεί κάποιες υποχρώσεις ε, και από τις πλευρές ε, και από τη Βοσνία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το εξή. Ε, πριν από τρεις μήνες πήγα στη Βοσνία και έκτοτε υπάρχει πρόοδος υπάρχει πρόοδος νομοθετικής φύσεως, κάτι το οποίο ανέφερε η συγγήτρια. Υπάρχει ή μάλλον θεωρώ ότι ε, εφόσον υπάρχει πρόοδος θα πρέπει να του ενθαρρύνουμε. Η παρέμβασή μας ε, θα πρέπει να είναι θετική και πρέπει να ε, διαφυλαχθεί η ισορροπία. Έχω να κάνω δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Πολλοί και σχολιαστές και άλλοι λένε το εξής. Αυτά που θέλουμε εμείς ε, να επιβάλλουμε κατά κάποιον τρόπο είναι γραφειοκρατικές ε, απόψεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως ε, να εξηγήσουμε στους πολιτικούς και στους πολίτες της Βοσνίας Ερσεγοβίνης ότι οι προτάσεις αυτές που καταθέτουμε είναι προς όφελος των ίδιων των κατοίκων της χώρας αυτής. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δικαστικό σύστημα. Αυτό όμως είναι προς δικό τους όφελος και όχι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό είναι λέει, το πρόβλημα των πολιτών. Έχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε ότι είναι σημαντικό να έχουν μια εύρυθμα λειτουργούσα δημοκρατία, μια δίκαιη δικαιοσύνη και αυτό για το δικό τους καλό, όχι για αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και αν τελικά πρόκειται να έχουμε ακόμα πιο στενές σχέσεις με τη χώρα αυτή, ε, θα πρέπει να σημειώσει κάποιες βελτιώσεις για να αναδειχθεί υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα για να βελτιώσουμε τις ε, σχέσεις ε, με τη χώρα αυτή και οι πολίτες και η χώρα το περιμένει αυτό. Όπως σας είπα όμως, αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να κατανοήσουν ότι αν ακολουθήσουν το σωστό δρόμο, πράγματι κάποια μέρα θα μπορέσουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Μπέλντα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η συγκήτρια, η συνάδελφος ε, κυρία Πάκα, σε εσά απευθύνομαι. Θέλω να σας πω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την πρόταση ψηφίσματος που καταθέσατε. Θα θυμάστε ότι πριν από κάποια χρόνια ε, είχαμε στην Ολομέλεια μια συζήτηση ε, για τον Ισλαμισμό, για τον Σαλαφισμό, δηλαδή για τις, τον Ισλαμικό ζηλωτισμό στην Βοσνία Ερσεγοβίνη. Πριν από λίγους μήνες ε, το περιοδικό Focus ε, στη Γερμανία προειδοποίησε και πάλι για την έξαρση του φανατισμού. Πρόσφατα μίλησα και με έναν ε, πυρογνώμονα που γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή Τούσλα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω τι ακριβώς πιστεύετε για τον επίσκοπο του Σεράγιβο. Εγώ είμαι ε, διαμαρτυρόμενος και ο επίσκοπος του Σαραγεύου είπε ότι αν ο φανατισμός αυτός, ο σαλαφισμός επεκταθεί στη Βοσνία Ερσεγοβίνη, το πρώτο θύμα θα είναι η φιλελεύθερη Βόσνοι. Εσείς τι πιστεύετε για την, αυτή την εξέλιξη του θρησκευτικού φανατισμού στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ προσωπικά Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει βέβαια να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια. Ε, δεν πιστεύω ότι ε, υπάρχει κάποιος ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να είναι περισσότερο αφοσιωμένος στο θέμα της Βοσνίας Αρζεγοβίνης από την εισηγήτρια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειες που καταβάλει και την καλή της θέληση. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Η Βοσνία Ερσεγοβίνη βεβαίως από στρατηγικής απόψεως ε, και κάτω από το πρίσμα της ε, πολιτιστικής ε, ολοκλήρωσης της ευρύτερης περιοχής είναι μια πολύ σημαντική χώρα και ποτέ δεν πρέπει να πάψουμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Βοσνίας Ερσεγοβίνης. Βέβαια, οι αρνητικές εξελίξεις δυστυχώς ε, υπερέχουν των θετικών. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι όσον αφορά την συμφωνία των πολιτικών κομμάτων για τη δημιουργία νέας κυβέρνησης και για την εκλογή Προέδρου και Πρωθυπουργού, αυτά τα εκλαμβάνουμε σε ένα θετικό μήνυμα. Αυτά πράγματι είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ε, προς ένα νέο ρυθμό εξελίξεων στη Βοσνία Σεχοβίνη. Επίσης, πιστεύω ότι ο διορισμός του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, του κ. Σόρενσεν, ε, είναι θετικό, ιδιαίτερα θετικό. και πρόσφατα ε, κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ αυτών και εγώ είχαμε ε, κάποια συνάντηση μαζί του και του εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του. Υπάρχουν βέβαια αρκετά πράγματα στη Βοσνία Σεγοβίνη τα οποία μας ανησυχούν. Εκτός από το πρόβλημα το οποίο ανέφερε μόλις τώρα ο κύριος Μπέλντερ, εγώ προσωπικά ανησυχώ όσον αφορά ε, δείγματα διχασμού στους νέους, τα οποία βέβαια αποτελούν, το αποτέλεσμα είναι απόρρια της ε, τεχνητής, του τεχνητού ορισμού συνόρων στη Βοσνία Ερσεγοβίνη μετά τον πόλεμο. Είναι απαράδεκτο τα παιδιά να μπαίνουν στο σχολείο από διαφορετικές πόρτες ανάλογα με την εθνικότητά τους. Από άλλη πόρτα μπαίνουν τα παιδιά των Σέρβων, από άλλη των Κροατών, αλλού πάλι των Μουσουλμάνων. Αυτά πράγματι είναι ε, ορατά προβλήματα στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Θα ήθελα κλείνοντας να πω το εξής. Είναι σημαντικό η κυβέρνηση της Βοσνίας Ερσεγοβίνης να αισθάνεται ότι χαίρει εκτίμησης και σεβασμού ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Πακ, έχετε το λόγο. Συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που ελέγχθησαν. Βέβαια, μόνο μία ερώτηση μου ετέθη. Το θέμα των ε, φανατικών ε, θρησκευόμενων στη Βοσνία Ερτσεχοβίνη. Ο κ. Μπέλτερ έχει δίκιο. Είχε προειδοποιήσει και παλαιότερα για αυτή την εξέλιξη. Αλλά αυτά τα πράγματα έχουν ε, προχωρήσει. Είναι η Βαχαμπίτσα από τη Σαντική Αραβία, οι οποίοι ε, προβαίνουν ε, σε ανοσιουργήματα και οι νέοι Βέβαια, τα θύματα που δεν έχουν δουλειά, αυτοί πέφτουν στην παγίδα των Μπαχαμπίτσι, οι οποίοι τους ε, προσλαμβάνουν ως ε, μισθοφόρου, αν θέλετε και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη μουσουλμανική κοινότητα ε, γιατί δημιουργείται κακή φήμη για αυτούς εφόσον πρόκειται για μουσουλμάνους. Έχετε δίκιο κύριε Μπέλτερ, θα έλεγα να καταθέσετε μία τροπολογία. Εγώ δεν το θίγω το θέμα στην έκθεσή μου, γνωρίζω πολύ καλά τον κίνδυνο. Εκείνο όμω το οποίο με εκνευρίζει ιδιαίτερα στην όλη υπόθεση είναι ότι ο επικεφαλής των μουσουλμάνων στην Βοσνία Ερσεχοβίνη, ο κύριος Τσέριτς, ο άνθρωπος αυτός ε, δεν αντιμετωπίζει στεναρά τους Βαχαμπίτς. Σε τελική ανάλυση είναι προς ε, όφελος ε, των δικών του των συνανθρώπων μουσουλμάνων να αντιμετωπιστούν στεναρά οι Βαχαμπίτς. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι τελικά οι Βαχαμπίτς πώς μπαίνουν στη χώρα αυτή. Δηλαδή αν εμείς ε, στις αρχές δεκαετίας 90 είχαμε ασχοληθεί περισσότερο με την Βοσνία Ερσεγοβίνη, κανείς δεν θα τους είχε καλέσει να έρθουν από Σαουδική Αραβία. Βλέπετε λοιπόν, τώρα πληρώνουμε τα λάθη της δεκαετίας του 90 και γι' αυτό το λόγο ακριβώς επειδή έχουν έτσι τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού το πρόβλημα. σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να δει κανείς πώς μπορεί να, να ανακαλέσει. Ε, αλλά ε, ε, ε, πριν από 10 χρόνια ήταν παρεμφερείς οι εκθέσεις και δεν βλέπουμε να έχει γίνει ουσιαστική έκθεση ουσιαστική πρόοδος δηλαδή πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε ε, αν μπορεί να γίνει ανάκληση διότι η δέσμευση για την, ε, ε, για την προσχώρηση υπάρχει από τη Θεσσαλονίκη και αν δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο κάποια στιγμή μπορεί να την επικαλεστούν. Λοιπόν, θα ευχαριστώ την κυρία Πακ. Πότε πρόκειται να ψηφίσουμε 7 1η Μαρτίου. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να καταλήξουν σε μια κοινή θέση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μεγάλη ε, πλειοψηφία. Ερχόμαστε στο 4, ένα ευαίσθητο θέμα. Το πρόσθετο πρωτόκολλο ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ισραήλ. Το οποίο επί πολλά χρόνια ήταν μπλοκαρισμένο ε, τώρα έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρέπει ε, να το προωθήσουμε η κυρία Ντεκάιζερ έχει καταρτήσει μία γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ίτερ και την παρακαλώ να μας παρουσιάσει τις θέσεις της. Κυρία Ντεκάιζερ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα και όπως είπατε ήταν ένα θέμα που είχε, είχε παραμείνει μπλοκαρισμένο επί σειρά ετών. Περιμένω 30 δευτερόλεπτα και συνεχίζω. Θέλω να υπενθυμίσω προτού προχωρήσω και εντοπίσω τα προβλήματα που διαπιστώνω να σας πω ποια είναι τα όρια του εγγράφου το οποίο έχετε μπροστά σας. Δεν είναι ακόμη ούτε ε, ψήφισμα ούτε γνωμοδότηση αλλά ένα έγγραφο εργασίας το οποίο καταγράφει τα σημεία τα πιο ευαίσθητα κατά την προσωπική μου γνώμη και τις, ε, τα ερωτηματικά που έχω σχετικά με μια τέτοια συμφωνία. Το πρωτόκολλο αυτό, το επιπρόσθετο πρωτόκολλο εις ε, την ε, Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ισραήλ ήταν μέρος του πακέτου το, αυτό το οποίο είχαμε ονομάσει upgrading, αναβάθμιση το 2008. Μπορεί όμως τώρα σήμερα να ολοκληρωθεί, να κυρωθεί χωρίς να θεωρηθεί πραγματική αναβάθμιση. Δηλαδή, στην κατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ισραήλ τεχνικά δεν πρόκειται για μια πραγματική αναβάθμιση. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που είχα και εγώ και μου εδόθησαν απαντήσεις και μάλιστα γραπτές από το, από γραφείο της κυρίας Άστον σχετικά με το θέμα αυτό. Δεύτερον, τι είναι μια συμφωνία ή ένα πρωτόκολλο που αναφέρεται αποκλειστικά στο Ισραήλ. Ε, ναι, αλλά πρόκειται για ένα, μια γενική συμφωνία η οποία θα μπορούσε να αναφερθεί σε όλες τις χώρες με τις οποίες υπάρχει πολιτική γυτνιάσεως και που σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο και οι οποίες θα μπορούσαν να προσχωρήσουν με απλοποιημένες διαδικασίες στην ευρωπαϊκή αγορά και αντιστρόφως. Είναι δηλαδή απλώς απλοποίηση της συμφωνίας. Οπότε το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα η οποία ε, τάχθη πέρα αυτές της συμφωνίας που χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια γιατί είναι η ολοκλήρωση του κοινοτικού κεκτημένου ε, επέλεξε έναν συγκεκριμένο τομέα στον οποίο είναι πολύ ισχυρό ε, το Ισραήλ δηλαδή τη φαρμακοβιομηχανία και είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους ε, παραγωγούς φαρμάκων διεθνώς. Είναι δηλαδή ένα τομέα στο οποίο η χώρα αυτή είναι πάρα πολύ ισχυρή. Όταν λοιπόν δούμε όλο το πακέτο και το εξετάζουμε, ε, λέμε ότι ίσως θα μπορούσε να τσουλήσει μόνο του. Αλλά υπάρχουν δύο ερωτηματικά τα οποία είναι σοβαρά. Ε, πρόκειται για νομικά ερωτήματα και τα νομικά ερωτήματα αναφέρονται στις πτυχές εδαφικότητος της συμφωνίας, δηλαδή την αναγνώριση των προϊόντων αυτών που θα πρέπει να γίνει βάση ε, μίας ε, βάσεως και το λέω άσχημα ε, αλλά ε, ουσιαστικά να γίνει κρυφίος κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή το Ισραήλ ε, θα καθορίσει το έδαφος επί του οποίου θα ισχύσει αυτή η συμφωνία που μπορεί να μην περιλαμβάνει τις απικίες, τους απίκους και ε, να υπάρξει μία διευκρίνηση ότι αυτά τα εδάφη τα οποία εμείς σαν Ευρωπαίοι θεωρούμε ε, σαν ε, εδάφη στα πλαίσια του εδάφους του Ισραήλ και όχι η Ισραηλινή νομοθεσία θεωρεί σαν εθνικό έδαφος και εδώ τοποθετείται και το θέμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Ε, δηλαδή, εδώ ε, δεν περιλαμβάνεται αυτούσια αυτό που θα έπρεπε να θεσπίζεται ε, και να ισχύσει και από πλευράς διεθνούς δικαίου και από πλευράς Ισραηλινού δικαίου. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι κάτι που δεν μπορώ να λύσω εγώ. Σας παρακαλώ λοιπόν κύριε ε, Πρόεδρε να ζητήσουμε μία νομική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Έχω δει την, επιτροπή, την απόφαση της Επιτροπής που εργάστηκε επί του θέματος πολύ σκληρά, αλλά η Επιτροπή μου λέγει ότι έχουμε ένα άρθρο το οποίο αντιλέγει ότι και ούτω καθεξής, αλλά εγώ θα ήθελα μία επίσημη θέση του Κοινοβουλίου. Εάν κάποιος μου πει ότι είναι μία προσπάθεια για να κερδίσω χρόνο Κύριε Πρόεδρε, δεν ε, έχω καμία πρόθεση να καθυστερήσω αυτό το φάκελο που είχε μπλοκαριστεί επί πολύ καιρό. Έφτασε η ώρα να τον μελετήσουμε, αλλά με ασφάλεια τόσο από νομική πλευρά όσο και από πολιτική πλευρά. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να υποβάλω σαν ερωτηματικό και προβληματισμό και είναι πολύ πιο σημαντικό παρόλο που το πρώτο δεν είναι πουσιώδες αλλά για τη δικιά μας επιτροπή είναι βασική η πολιτική σκοπιά και σκοπιμότητα. Δηλαδή έφτασε η στιγμή, έχει φτάσει η στιγμή να ε, συνάψουμε αυτή τη συμφωνία ακόμη και αν τεχνικά δεν πρόκειται για μία αναβάθμιση. Εδώ υπάρχει μία σειρά από επιχειρήματα τα οποία ανέφερα απλώς στο έγγραφο εργασίας και είμαι διαθέσιμη για να απτύξω περαιτέρω στην επόμενη διατύπωση Καταρχήν δηλαδή τη συνεκτικότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της εφαρμογής των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα διάφορα ε, έγγραφα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, οι χώρες με τις οποίες συνάπτουμε συμφωνίες θα πρέπει να, είναι, να σέβονται πλήρως το διεθνές δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο και ως εκεί πάμε καλά. Αλλά έχουμε τη την συνήθεια επειδή ε, συνάπτουμε συμφωνίες με χώρες οι οποίες δεν είναι άμεμπτες από πλευρές ανθρωπίνων δικαιωμάτων να θεωρούμε ότι δεν κοιτάμε το κράτος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τις τάσεις. Αν η κατάσταση βελτιώνεται ή επιδεινώνεται. Πιστεύω λοιπόν ότι από αυτή τη σκοπιά, όταν αναφέρομαι στην ε, συνοπτική παρουσίαση που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συμβούλιο της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ισραήλ του Φεβρουαρίου 2011, δηλαδή προενός έτους, ε, υπήρξε ένα συμβούλιο που διεξήχθη και όπου είχαν ε, ε, επισημανθεί διάφορα προβλήματα τα οποία ήταν ε, σοκαριστικά ενοχλιστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ελέγεται καταδικάζουμε, λυπούμεθα, θα διαπιστώνουμε με λύπη και δεν αναφέρομαι εδώ σε όλες τις εκθέσεις οι οποίες έχουν ε, δημοσιευθεί από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που επισημαίνουν διάφορα προβλήματα. Εμείς στο Συμβούλιο εκείνο λυπούμεθα για τη ε, συνέχιση της πολιτικής απίκων που είναι μία σαφής απειλή για την ειρήνη ήμασταν ε, ε, αντίθετοι εις ε, την περικύκλωση της και αποκλεισμό της Γάζας και λέγαμε, ζητούσαμε άρση του αποκλεισμού και τα μέτρα που λαμβάνονταν θεωρούσαμε ότι ήταν ανεπαρκή. Λυπούμεθα για τη στάση των Ισραηλινών αρχών και ανησυχούμε πάρα πολύ για το την νομοθεσία σχετικά με τις ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Αναφέρουμε λοιπόν στα τέσσερα αυτά σημεία και όταν σήμερα ένα χρόνο μετά ε, εξετάσω πού βρισκόμαστε σε σχέση με το τότε κείμενό μας βλέπουμε ότι το πρόβλημα των απίκων έχει εξελιχθεί αλλά προς την λανθασμένη κατεύθυνση. Δηλαδή, τη στιγμή όπου στον ΟΗΕ ο πρόεδρος Αμπάς ζήτησε ε, να ε, γίνει αποδεκτός το κουαρτέτο κατήρτισε αυθημερών ε, ένα χάρτη πορείας και είπε ότι αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι να εισαχθεί η, η, Παλαιστίνη στον ΟΗΕ αλλά να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί η ειρήνευση και αυτό το οποίο εμπόδιζε ήταν η συνέχιση των απίκων Έπρεπε λοιπόν να καθοριστούν τα κριτήρια επί των οποίων ε, θα ε, καθορίζονταν τα σημεία προς διαπραγμάτευση. Η καταληκτική ημερομηνία ε, ήταν 27 πρώτου, δεν έγινε τίποτα και τώρα διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση δεν εξελίσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση και δυστυχώς είμαστε αποτελματωμένοι στην ίδια κατάσταση που είμαστε και πριν ένα χρόνο. Γι' αυτό και λέω κύριε Πρόεδρε ότι το σήμα που μπορεί να δώσει το, η Επιτροπή μας δίδοντας τώρα μία θετική συμφωνία ε, σε, ε, αυτή την, ε, σε αυτό το πρωτόκολλο ακόμη κι αν μιλάμε για τη φαρμακοβιομηχανία μόνο είναι όμως μία πολιτική κίνηση η οποία μου φέρνεται σαν μία ένδειξη ότι ασχέτως του ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε όπως είχαμε ε, διακηρύξει στην ε, έκθεσή μας ή στην έκθεση της Μαρία Ακτιβιέ ε, ότι θα το χρησιμοποιήσουμε σαν μέσο για να έχουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή δίνουμε κάτι για να έχουμε κάτι καλύτερο. Εγώ αυτό που περιμένω είναι μια βελτίωση επιτόπου και ε, μία κίνηση στο θέμα των απίκων, τους οποίους ποτέ δεν αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα πολιτικά επιχειρήματα τα οποία έχω. Όσον αφορά την, ε, τα νομικά επιχειρήματα, Πιστεύω ότι ε, υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα, δεν είναι ε, μία προσπάθεια να καθυστερήσω το θέμα. Θα ήθελα όμως η ε, νομική υπηρεσία να με διαβεβαιώσει ότι αυτή η συμφωνία είναι βιώσιμη πολιτικά, πράγμα με το οποίο διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ως πρώτος ο μιλητής, ο κύριος Πίτερλε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Πίτερλε. Η αλήθεια είναι ότι την προξενή έκπληξη το ότι αυτό το επισυνοπτόμενο πρωτόκολλο εκκρεμούσε ή και ίσχυε τόσο καιρό. Τώρα λοιπόν, ρίχνοντας μια ματιά στο κείμενο, αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τις διαπραγματεύσεις έχοντας κατά νου μόνο το δικό τη συμφέρον. Και επομένω προσφέρει μια, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το δικο της συμφερον Έχει εδώ κάποιε τεχνοκρατικέ διατάξει όσον αφορά την συνεργασία σε συγκεκριμένου τομεί. Δεν ε, περιλαμβάνει κάποιο είδου ε, αναβάθμιση όσον αφορά το τι ισχύει για τη χώρα. Το Ισραήλ επίση έχει προωθήσει κάποιε μεταρρυθμίσει όσον αφορά την εθνική νομοθεσία και αυτό το έκανε ε, λαμβάνοντα υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο και επίση τι ε, συμφωνίε συνεργασία. Ε, συμφωνώ, θεωρώ τέλο πάντων ότι το προηγουμένο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται επίσης να προβεί και σε σύνταξη νομικής γνωμοδότησης. Το θέμα είναι δύσκολο, είναι λεπτό. Οπότε και γι' αυτό ε, το μάλλον επιβάλλεται να υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση. Επίσης, εδώ είναι θέμα αρχών. Αυτό που είπε η κυρία Ντεκεζέρ, ότι δηλαδή έχουμε εδώ ένα εργαλείο, ένα μέσο πολιτικής, ούτως ώστε να επιδιωχθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Πρόκειται επομένω για πλαίσιο το οποίο ακριβώς καλύπτει κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Επομένως και εμείς θα πρώτο λάβουμε αυτό υπόψη για την τοποθέτησή μας. Θέμα αρχών επαναλαμβάνω. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ακριβώς προέβη, τι έλαβε υπόψη για αυτή την νομική γνωμοδότηση. Πάντως και για το Κοινοβούλιο και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να υπάρξει μια απεμπλοκή στην όλη κατάσταση και τελικά να εγκριθεί αυτό το σημαντικό μέσο πολιτικής και τόσο να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος, κύριος Σας ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θα έρχομαι να συμφωνήσω με αυτή την πρόταση ότι δηλαδή θα πρέπει να απευθυνθούμε για να λάβουμε μια νομική γνωμοδότηση. Όμως, εδώ το θέμα παρουσιάζει ένα πρόβλημα. Τι θα θεωρούμε εδώ πέρα, ότι είναι τεχνοκρατικό, ε, αυτή η συμφωνία ή θα πρέπει να τη βέβαια πλευρά πολιτική. Γιατί κάθε φορά, κάθε φορά ε, μπορεί το, το, το τεχνοκρατικό να χρησιμοποιείται για σκοπούς πολιτικής. Άρα θα πρέπει εδώ να αποφασίσουμε. Θα κάτσουμε και θα ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά το, το κειμένο ή θα πρέπει ακριβώς να το συζητήσουμε σαν να ήταν μέσω άσκησης πολιτικής. Βεβαίως και έχουμε αποκρισταλώσει κάποια άποψη και ότι θα πρέπει την άλλη μεριά να τοποθετηθούμε τελικά θα πρέπει κάπως να, να δείξουν προς τα έξω στους εμπλεκομένους ότι θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν όμως. Το πρόβλημα είναι ότι με αυτήν την, την, την αναβάθμιση που είχε παγώσει τόσο καιρό εδώ, ε, τα μέρη δεν προχωρούσαν στις διαπραγματεύσεις και τελικά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και κάποιες δεύτερες σκέψεις ε, και κίνητρα ε, κάποια πιστοβουλία τέλο πάντων από πλευρά των εμπλεκομένων οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τι μεταβλητέ για να καταλήξουμε στο πώ θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τελευταίο, το οποίο νομίζω θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και βεβαίω δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με το ότι πρέπει να αναζητήσουμε κάποια γνωμοδότηση. Όταν μιλούμε για κράτο για επικράτεια του Ισραήλ, τι, τι γίνεται. Αμφισβητούμε τα πάντα σε σχέση με την οντότητα του κράτου. Πάσα συμφωνία με το Ισραήλ θα πρέπει να περνάει μέσα από αυτό το, το πρόβλημα ε, της επικρατείας. Επομένως αυτό σημαίνει ότι ευθύ εξ αρχής δυναμητίζουμε ε, τις σχέσεις μας με ένα πάρα πολύ σημαντικό κράτος. Επομένως ε, εμείς ως Επιτροπή δεν θα πρέπει να δίνουμε αυτή την εντύπωση ότι δηλαδή με ερωληπτούμε υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Ευχαριστώ. Κύριε Γιαννάκο. Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε ήδη κάνει μία συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής εν και τοποθετήθηκα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έναντι της πρότασης της κυρίας Ντεκάιζερ να ζητηθεί νομική γνωμοδότηση αρνητικά. Δεν είναι δυνατόν μία πολιτική και τεχνική υπόθεση να χρειάζεται μία νομική γνωμοδότηση όταν έχει αποφανθεί το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι χρέος της εισηγήτριας είναι να κάνει την εισηγησή της. Μπορεί η εισηγησή της να είναι αρνητική. Είναι δικαίωμά της να κάνει αρνητική εισήγηση αλλά δεν νομίζω ότι η Επιτροπή μας έχει το δικαίωμα να καθυστερεί σκόπιμα μία εισήγηση προκειμένου να μην δώσει τη γνώμη, τη της σε μια άλλη επιτροπή και δεν νομίζω πως η αρμόδια επιτροπή θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο για να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει βέβαια τις παραμέτρους, τις πολιτικές, δηλαδή το Παλαιστινιακό ζήτημα, τη σύγκρουση, τη Γάζα και όλα τα σχετικά. Ε, αλλά κύριε Πρόεδρε, εάν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαβεβαιώσει ότι δεν συναλλάσσεται με κανέναν ο οποίος έχει παρόμοια προβλήματα, τότε να το κάνουμε και γι' αυτό. Αυτό όμως δεν συμβαίνει όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να εκθιάσω πλέον εκτίματα αυτής της σύμβασης. Είναι γεγονός ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα του Ισραήλ είναι αρκετά υψηλής ποιότητας και εξ όσων γνωρίζω και χαμηλής τιμής. Αλλά δεν θα μπω στην ουσία αυτής της υπόθεσης. Η δική μας άποψη είναι ότι είναι σοβαρό λάθος να αναζητούμε νομικές γνωμοδοτήσεις επί ενός πολιτικού θέματος και ότι καλείται η συγγήτρια να αντιμετωπίσει το ζήτημα ως συγγήτρια κάνοντας τη γνωμοδότησή της και Ας κάνει αρνητική γνωμοδότηση. Εδώ είναι η Επιτροπή Εξωτερικών να αποφασίσει με πλειοψηφία όπως αποφασίζουν όλα τα κοινοβούλια αλλά το να βρίσκουμε δικαιολογίες στέλνοντας την υπόθεση αυτή ε, στην, ε, είτε στην νομική επιτροπή του κοινοβουλίου είτε στην νομική υπηρεσία του κοινοβουλίου αυτό αποτελεί απλώς κολυσιεργία πολύ περισσότερο κύριε Πρόεδρε που δεν θα λύσουμε εμείς εδώ την σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης δηλαδή επί της ουσίας είναι προφανές ότι δεν υπάρχει επιθυμία να γίνει αυτή η γνωμοδότηση. Λοιπόν, εγώ επιμένω εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι η συγκήτρια οφείλει να έχει μια γνωμοδότηση και ας είναι αρνητική και να τη φέρει στην Επιτροπή να αποφασίσουμε χωρίς περιττές κολυσιεργίες και χωρίς υπερβολές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Äh, äh, πολύ ωραία. Το λόγο έχει η κυρία Νίλσεν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Νομίζω ότι η κυρία Ντεκεζέρα έχει δίκιο όταν ε, ζητεί να δοθεί αυτή η γνωμοδότηση. Και εγώ είμαι πέρα ε, του να το ζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως τα προανέφερε η συνάδελφος. Ένα τεχνικό, τεχνοκρατικό θέμα, ας πούμε τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία τώρα ε, παρασκευάζονται στο Μαλέι, ε, εκεί κοντά στην Ιερουσαλήμ που είναι ένας επικισμός. Ε, οπότε έχουμε εκεί αυτή την φαρμακοβιομηχανία στην πούμε που είναι εγκατεστημένη ή στα κατεχόμενα. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για να θεωρήσουμε ότι είναι τεχνικό, τεχνοκρατικό το ζήτημα. Εγώ επίση θέλω να σα αναφέρω κάτι για μια κοινοβουλευτική έκθεση η οποία παρουσιάστηκε στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση από λίγε εβδομάδε και που αφαιρούσε το ζήτημα ε, των υδάτων, του ύδατο τέλο πάντων στην, στην, Παλαιστίνη. Αυτό το οποίο χρησιμοποιείται για βιομηχανικού φαρμακευτικούς σκοπούς. Θα πρέπει να λέτε ότι έχουμε 450.000 ε, ε, επίκους στην Περιορδανία οι οποίοι ε, καταναλώνουν πολύ περισσότερο νερό από ότι τα 2,5-2 εκατομμύρια 300 Παλαιστίνοι. Επομένως η χρήση του ύδατος εδώ αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα. Η δε βιομηχανία βεβαίως καταναλώνει νερό. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι δεν συνδέεται το, το, το, το, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το τεχνικό αυτό θέμα του ύδατος. Επομένως θα πρέπει και θα οφείλουμε τα ανθρωπινά δικαιώματα να ενταχθούν ε, στην καρδιά της πολιτικής μας και οπότε να λάβουμε υπόψη αυτό το κείμενο ε, γιατί εκεί περιέχονται και θίγονται όλα τα σημαντικά ζητήματα τα οποία δικαιώνουν το να μην συνεχίσουμε προς την ίδια ρότα. Και οπότε τον Ιούλιο 2011 έχουμε τους 27 επικεφαλείς των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στην Ιερουσαλήμ ε, ενδεικτικά είχαν απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της είπανε ότι θα πρέπει να βρει ένα νομικό μέσο και να, να, να, να ε, πάσα ευρωπαϊκή επένδυση στους επικισμούς. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, δεν μπορούμε να, να λέμε ότι αλλού είναι τα πολιτικά, αλλού είναι τα τεχνικά και κυρίως να, να, να, να παραβλέπουμε τα θέματα διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά και το νομικό θέμα εδώ είναι αυθεντικό. Είναι νόμιμο, είναι σύνομο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκεί εμπορία με κάποια χώρα η οποία κατέχει μια επικράτεια και εκμεταλλεύεται με καταχρηστικό τρόπο, περιβολικό, τους εκεί κατοίκους και εμείς να ανασιωπούμε και όλα αυτά να αντιβαίνουν κατάφορα εις την συνθήκη της Γενέβης. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τους συναδέλφους να είναι λίγο πιο σύντομοι κατά τρόπον ώστε να μην ε, χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση για να συζητήσουμε όλο το θέμα της Μέσης Ανατολής. Ο κύριος Τάνοκ. Πρόεδρε, για να σας πω και να παραπονεθώ ότι μου δώσαν τα κείμενα μόνο στα γαλλικά. Τι γίνεται εδώ, παρελκυστική τακτική είναι αυτή σε σχέση με το τι θα κάνουμε για το κείμενο του Kaiser. Γιατί ρώτησα τον Ολλανδό συνάδελφο και μου αυτός πήρε τα αγγλικά. Εγώ λοιπόν πήρα τα γαλλικά, το οποίο θα, θα με καθυστερήσει μέχρι να καταλάβω περί των πρόκειται. Πάντως εγώ συμφωνώ με το ΕΛΚ ε, ότι είναι καθήκον μας να πάψουμε αυτές τις παλιστικές τακτικές, ε, αυτό τράβηξε δύο χρόνια. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια γνώμη και να μην λέμε άντε ας ψάξουμε τη γνώμη των νομικών, να ανακατεύουμε τα διάφορα άσχετα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την τεχνική έκθεση για ένα θέμα εμπορικό μεταξύ μιας δημοκρατίας του Ισραήλ, με την οποία έχουμε αγαστές πολιτικές και σχέσεις. Και από την άλλη μεριά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν αυτού νομίζω ότι έχουμε ως συνέπεια το ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εξαιρετικά παγκοσμίου φήμης Ισραηλινά φάρμακα. Άρα με όλα αυτά παραβλάπτουμε τους δικούς μας συμπολίτες κυρία Ντεκάιζερ πρεσβεύει ότι δεν ενεργούμε σύνομα σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι τελείω άλλο ζήτημα όσον αφορά το Ισραήλ, όσον αφορά την ε, εδαφική ακεραιότητα, ε, τι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι άσχετο θέμα. Εμεί εδώ θα πρέπει να ζυγίσουμε πέρα και τα κατά αυτή τη τεχνική συμφωνία, να δούμε τι γίνεται με αυτά τα, τα βιομηχανικά προϊόντα. Ε, δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε στο Μεσανατολικό αντί να συζητούμε το συγκεκριμένο. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να σταθμίσουμε το πώ θα βρούμε βεβαίω μια λύση, τόσο να υπάρχει ασφάλεια, διμερία στην περιοχή. Όλα αυτά σύμφωνοι. Όμω δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συνεχώ ε, φρένο σε κάθε συζήτηση, όπω εδώ στο συγκεκριμένο θέμα για τι εξαγωγέ των φαρμάκων. Δεν βοηθάει καθόλου. Οπότε παρακαλώ και η Επιτροπή μα και το Κοινοβούλιο γενικότερα να τοποθετηθεί επί τη ουσία για αυτήν την τεχνική συμφωνία. Να ψηφίσουμε, να μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη κανονικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλντερ. Θα είμαι πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνο. 100% με τον κύριο Τάνοκ. Και παρακαλώ. Ο εισηγητής, η εισηγήτρια, να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια άποψη. Είμαστε κοινοβούλιο. Αυτό είναι η δουλειά μας. Πρόεδρος. Είναι το λόγο στον επόμενο. Ευχαριστούμε την κυρία Ντεκάιζερ για το έγγραφο. Από τότε που ήταν συντονίστη των σοσιαλιστών είχαμε αγαστές σχέσεις με την κυρία Ντεκάιζερ όμως επί του προκειμένου νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύστοχα τα οποία μας λέει. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλουμε είναι το πώς, όπως προβλέπετε, θα υπάρχει μια γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτή την εμπορική συμφωνία Ένωσης Ισραήλ. Αυτό το οποίο επομένω πρέπει να κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας είναι να προχωρήσουμε σε μια έκθεση. Οι 27 υπέραψαν τη συμφωνία και κατόπιν δύο χρόνια ε, κόλλησε το θέμα. Και λέμε τώρα για γνωμοδότηση. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει ο Ντεκάιζερ είναι πολιτικά φορτισμένα. Δικαιούται να το κάνει κάτι τέτοιο. Όμως εδώ έχουμε την κύρωση τεχνικής συμφωνίας. Έχουμε φυσικά τα πολιτικά θέματα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του από τη διαδικασία ερήνευσης στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Όμως, τροχοπέδι δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως ε, έχετε σαφώ κύριε Γκάζο και συμφωνούμε ούτω ή άλλω σε πολλά σημεία. Όμω, επί του προκειμένου, θα πρέπει εμεί να εκδώσουμε, να προχωρήσουμε στην, στην ολοκλήρωση τη έκθεση τη γνωμοδότηση. Αυτό κύριε Ντεκάιζερ δεν είναι έγγραφο εργασία. Είναι δήλωση πολιτικών πεπιθήσεων. Να μα λέτε ότι δεν έχουν οριμάσει πολιτικέ συνθήκε. Εντάξει, ε, τι μπορείτε να τι ε, προωθείτε. Όμω πρόκειται εδώ για μια χωριστή διαδικασία. Διαφορετική από αυτά τα οποία προβλέπονται. Και μιλούμε για τεχνικό θέμα που δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να φρενάρεται από την πάλι στην Ισραηλινή διαμάχη έχουμε εδώ πέρα μία ε, μία ανάγκη γνωμοδότησης και άρα θα πρέπει σε σχέση με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας να αποφανθούμε. ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην έψω αυτή, στην Επιτροπή, βρισκόμαστε για να αναπτύσσουμε τα όνειρα, τα όραματά μας και έτσι να διαμορφώνουμε την κοινή άποψη. Βεβαίω και είμαστε υπέρ της ειρήνη στη Μέση και είμαστε κατά της ε, βίας, του πολέμου. Θέλουμε όμως να πρετανεύσει η ειρήνη εκεί και αυτό προς όφελος ε, και του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Και εγώ θα ήθελα να υπάρχει επάρκεια ύδατος και θα ήθελα να υπάρχει δίκη ε, κατανομή των υδάτινων πόρων. Όμως, σήμερα οφείλουμε να τοποθετηθούμε επί του προκειμένου. Δεν θα αλλάξουμε σήμερα τον κόσμο. Τίποτα από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένω δεν θα αλλάξουν ε, την, την, την κατάσταση Μέση Ανατολή. Όντω, ε, με κάθε σεβασμό ακούω τα όνειρα τη κ. Ντεκάιζερ, διότι δίνει μάχη για κάποιε αξίε. Όμω, θα πρέπει εμεί να αναρωτηθούμε κατά πόσον η τοποθέτησή μα θα βοηθήσει να επιληθεί το πρόβλημα. Είμαστε υπέρ κατά τη κύρωση αυτή τη διεθνού συμφωνία. Επομένω, νομίζω ότι αν απευθυνθούμε στην νομική υπηρεσία για γνωμοδότηση, δεν πρόκειται αυτό να βοηθήσει καθόλου στο να βρεθεί κάποια λύση στο Μεσανατολικό, διότι όλα αυτά τα οποία είπε η συγγήτρια, όλα τα, τα εδαφικά προβλήματα είναι γνωστά. Έτσι κι αλλιώς, σε όλα τα προϊόντα αναφέρουν που έχουν κατασκευαστεί αυτό και το κάνει το Ισραήλ. Οπότε βεβαίως ε, το ότι δεν είναι καλή η πολιτική συγκυρία, το ότι υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή, αυτό ισχύει εδώ και 60 χρόνια και ίσω θα ισχύσει για άλλα τόσα. Επομένως, πού καταλήγουμε. Να μην κάνουμε τίποτα επειδή είναι έτσι η κατάσταση στην περιοχή. Άρα, εμεί δικαιούμεθα εναντί Κομισιόν, Συμβουλίου και των χωρών που θα ήθελαν να τεθεί σε σχημή συμφωνία, να δούμε κατά πόσον θα θέλαμε να, υπάρξει ή να μην υπάρξει μια τέτοια συμφωνία που δεν είναι πολιτική, είναι εμπορική. Εάν επομένω, εμείς εδώ και τώρα αρχίζουμε να συζητούμε για ανθρώπινα δικαιώματα, τότε τότε οι συμπολίτες μας, οι ψηφοφόροι μας θα γυρίσουν και θα μας πούν όμως εμείς θέλουμε να έχουμε προσβασιμότητα σε αυτά τα σημαντικά φάρμακα. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μα βοηθήσει να τα αποκτούμε πιο εύκολα αυτά. Εάν κάτσουμε λοιπόν και λάβουμε υπόψη όλε αυτέ τι επιφυλάξει και εμβολίε τη κυρία Ντεκεζέρ, εάν επομένω πούμε ότι α ε, λύσουμε τα αυτά προβλήματα πρώτα που θα... Αντίθετα, εάν τώρα λύσουμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ίσω αυτό βοηθήσει να λυθεί το ευρύτερο πολιτικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα περιοριστώ στο να σας πω ότι η συμφωνία αυτή έγινε βάσει συγκεκριμένης εντολής του Συμβουλίου να συνάπτουμε συμφωνίες αυτού του είδους με χώρες ε, ευρωμεσογειακές. Έχουμε λοιπόν ε, εμπλακεί σε τέτοιες διαπραγματεύσεις με μία σειρά κρατών. Το Ισραήλ είναι ίσως η πλέον αναπτυγμένη και η πλέον προοδευτική από πλευράς ε, ευθυγραμμίσεως και απευθυνθήκαμε σε αυτούς γιατί είχαν κάτι να μας προσφέρουν άμεσα. Δεν μπορώ να διαβεβαιώσω ότι εμείς θέλαμε να κάνουμε μία τεχνική συμφωνία για να βελτιώσουμε τις εμπορικές σχέσεις, ιδίως διότι το Ισραήλ είναι, το Ισραήλ είναι ε, ε, πολύ δυνατός παίκτη στη γεωργία και ε, είχαμε επισυνάψει μία ανάλυση πέραν των ρυθμιστικών θεμάτων και γι' αυτό θέλαμε η συμφωνία αυτή να επιτύχει μία κίνηση αντί για δύο. Και ε, είχαμε συμφωνήσει ότι αν δεχθούν τους ε, όρους μας θα δεχθούμε και εμείς τους όρους τους για να επιτρέψουμε ε, την πρόσβαση των προϊόντων τους στην αγορά μας. Ο στόχος ήταν να γίνει ένα τεχνικό έγγραφο το οποίο θα βελτίωνε τους, ε, ε, εμπορικούς, ε, τους όρους εμπορικής συναλλαγής. Βεβαίως όποτε καταρτίζεται ένα τέτοιο έγγραφο μπλέκεται η νομική υπηρεσία η οποία ήταν στο πλευρό μας καθ' όλες τις διαπραγματεύσεις και στο τέλος η συμφωνία ε, παραπέμφθηκε στην νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ε, ενεκρίθη οπότε το έγγραφο αυτό θεωρήσαμε ότι ε, θα περιλαμβανόταν ε, και εις ε, την εμβέλεια της συνθήκης της Λισαβόνας οπότε το ξανα εξέτασε και η δική μας νομική επιτροπή της, Ευρωπαϊκής, ε, της ε, Κομισιόν δηλαδή και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αρκετή λοιπόν βεβαιότητα στη γνώμη των ε, ομολόγων μας μπορούμε να πούμε ότι κατά τη γνώμη μας αυτή η συμφωνία συνάδει με την διεθνή νομοθεσία και με τις συνθήκες. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω και να επαναλάβω ότι πρόκειτο για ένα εμπορικό έγγραφο βάσει συγκεκριμένης εντολής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το θέμα της εδαφικής εφαρμογής. καλύπτεται στο τμήμα 4. Κοντά ε, στο 4α δεν χρειάζεται να ε, αναφερθώ εγώ διότι θα δείτε ότι αναφέρεται ή στην ε, εδαφική ε, εφαρμογή και ε, εφόσον υπάρχει εφαρμογή της βασικής συμφωνίας η οποία δεν έχει αλλάξει εδώ θα, ε, τα πρωτόκολλα θα ακολουθήσουν τη βασική συμφωνία αλλά όπως σας είπα στο τμήμα 4 ρήτρα 2 παράγραφος α το καλύπτουμε. Αυτό είναι μεγάλη ε, ε, πρόοδος και έχουμε την ε, ίδια άποψη. Οπότε αντιλαμβάνουμε ότι εφόσον έχουν ερωτηθεί τρεις νομικές υπηρεσίες οι οποίες ποτέ δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους έχουμε τρεις διαφορετικές απόψεις. Αλλά ε, είχα παρακαλέσει, το, είχα παραβλέψει τον κύριο Βάιγκελ και του δίνω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για... Είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Θα πρέπει εδώ να κάτσουμε να δούμε τις αποχρώσεις όλων των, των, των ε, απόψεων γιατί όντως εδώ πέρα έχουν πάρα πολλές οικονομικές σχέσεις και ε, ε, εντάξει, όλε οι σημαντικέ χώρε είναι σημαντικοί εταίροι μα. Όμω αυτή τη στιγμή, ε, όταν θέλουμε να συνάψουμε κάποιε εμπορικέ συμφωνίε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτέ οι εμπορικέ συμφωνίε δεν θα πρέπει να, να, τα εσκαμμένα, δηλαδή τι κόκκινε γραμμέ τη ε, διεθνού συνεργασία, τη εμπορική συνεργασία, τη οικονομική συνεργασία, όπω ισχύει διεθνώ. Οπότε, εάν θέλουμε εμεί να διαδραματίσουμε στη διεθνή σκηνή έναν ρόλο που να μην είναι απλά και σκέτα εμπορικό, θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Θεωρώ ότι η κυρία Δικαζέρ ε, αυτό ακριβώς ε, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όσον αφορά το πρόβλημα της έντασης που υπάρχει, της προστριβές στην Μέση Ανατολή, ε, ναι, θα πρέπει τελικά να δοθεί ειρηνική λύση. Επίσης, άλλο πρόβλημα. Το τι θα γίνει όσον αφορά αυτή την επέκταση την συνεχή επέκταση των επικισμών. Γιατί τη συγκεκριμένη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Τα είδαμε, τα διαπιστώσαμε στα πλαίσια του διαλόγου Μπανκιμούν Νετανιάχου. Έλεγε ο Μπανκιμούν ότι θα πρέπει να υπάρξει περιορισμό, να υπάρξει ένα φρενάρισμα σε αυτού του επικισμού και έλεγε ο Νετανιάχου όχι, ε, δεν είναι προγραμματεύσει αυτέ και εκεί υπήρχε η ρήξη. Επομένως, να διαπιστώσουμε ότι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ και αυτό το θέμα και όλα τα άλλα έχουν και πολιτικό χαρακτήρα γιατί έχουν σχέση με το Ισραήλ. Εμείς δε, ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε ευθύνη και αρμοδιότητα να ε, παίρνουμε το πράγμα όλες τις ε, απόψεις. Δηλαδή, να αναρωτηθούμε, θέλουμε ή δεν θέλουμε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να επιδεινωθεί η κατάσταση εκεί. Γι' αυτό σας λέω, ας λάβουμε υπόψη το κείμενο αυτό το οποίο συνδέει την εμπορική συμφωνία με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ακόμα με την εμπορία προϊόντων τα οποία κατασκευάζονται σε κατεχόμενα εκεί όπου όλος παρανόμος προβαίνει σε αυτές τις ε, ενέργειες των, των, τοπικών, των υδάτινων πόρων το Ισραήλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποβάλω μια πρόταση και στο τέλος ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ. Ε, πρώτον, θέλω να πω ότι πρέπει να τοποθετηθούμε. Είναι δυνατόν όσον αφορά στο Σύνταγμα να προηγηθεί η ε, Επιτροπή, αρμόδια Επιτροπή και να αποφασίσει. Και την περίπτωση αυτή θα μπορούν να αποφασίσουν χωρίς να λάβουν υπόψη στη δική μας την άποψη. Αυτό είναι ένα γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προτείνω, ανεξάρτητα με το τι θα κάνουμε τελικά, προτείνω κυρία Ντεκάιζερ να υποβάλλετε σχέδιο έκθεσης για να μην μείνουμε εκτός παιχνιδιού. Τώρα, ε, κατά πόσον θα εγκριθεί η έκθεση όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Καλύτερα όμως ε, να κατατεθεί σχέδιο έκθεσης ε, εκ μέρου της Επιτροπής. Εγώ έτσι φρονώ. Το δεύτερο είναι το εξής. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι την πολιτική ιεράρχηση. Η κυρία Ντεκάιζερ ανέφερε πολλές επιφυλάξεις και νομίζω σχεδόν όλοι συμφώνησαν με αυτές. Μόνο που τίθεται το εξής ερώτημα. Αυτό ή αυτά, οι επιφυλάξεις αυτές αποτελούν λόγο για να απορρίψουμε ένα πρόσθετο πρωτόκολλο ως παράρτημα μιας υπάρχουσας συμφωνίας. Και όπως είπε ο κ. αυτό σε τελική ανάλυση δεν είναι ένα πρωτόκολλο που θα αποβεί προς όφελός μας. Γιατί ε, αν απορριφθεί αυτό το πρωτόκολλο, ενδέχεται ε, το γεγονός αυτό να μην εκνευρίσει τόσο το Ισραήλ όσο εμάς. Νομίζω ότι πολλές φορές πρέπει κανείς να σκέφτεται και το θέμα της χρησιμότητας ε, όταν ε, καλείται κανείς ε, να αποφασίσει. Και κάτι άλλο το τελευταίο που το είπε και η Κομισιόν, ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που αφορά το σύνολο των κρατών της Μεσογείου. Δηλαδή, αν έχουμε προβλήματα με άλλα κράτη Euromed και πούμε ότι θα μπλοκάρουμε διότι το σχάριν ε, στην Αίγυπτο ε, αντιμετωπίζουν δικαστικές διαμάχες ή ΜΚΟ ή κάτι παρεμφερές. Μα αν γίνει αυτό τότε ποτέ θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε παρεμφερή θέματα γιατί και σε άλλα σημεία της ε, Ευρωμεσογείου δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουν επιβληθεί το κράτος δικαίου και η δημοκρατία ε, παρά τις τελευταίες εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, εγώ προτείνω κατά πόσον θα πρέπει η κυρία Ντεκάιζερ να σκεφτεί μαζί με την Ίντερ να προσπαθήσουμε να θεσπίσουμε ένα ψήφισμα και μέσα στο ψήφισμα αυτό να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας, κυρίως εκείνες που έχουν σχέση με τις ε, εδαφικές ε, εφαρμογές. Ίσως μπορούμε να δώσουμε εντολή στην Κομισιόν να εξετάσει αυτά τα θέματα και άλλα για να ε, βρούμε κάποια μέση οδό. Και μετά θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο, όπως σας είπα, για να μην παραγωνιστεί πλήρως η Επιτροπή μας. Σήμερα θα το προτείνω αυτό ε, στην συνάντηση των συντονιστών και βλέποντας ότι μετά από πίεση της ε, κυρίας Άστον οι δύο πλευρές ε, έχουν έρθει και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βλέποντας ότι τώρα πλέον σε πολιτική πλευρά σε πολιτικό επίπεδο έχει επέλθει κάποια συμφωνία Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο ε, στην Επιτροπή μας να γίνει μια διεξοδική συζήτηση. Είτε θα είναι ακρόαση αυτή είτε όχι. Θα μπορέσουμε όμως να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα τα οποία πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Ντεκάιζερ. Και μετά, η, το, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Ντεκάλια θα έχει τη σιγουριά ότι όλα αυτά δεν τα απορρίπτουμε, συνεχίζουμε να τα παρακολουθούμε. Αυτή είναι λοιπόν μια δυνατότητα να προχωρήσουμε με αυτό το πακέτο και πολιτικά θα επιτύχουμε αρκετά, θεωρώ, αλλά και από την άλλη πλευρά θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και όλα τα άλλα θέματα. Κυρία Ντεκάιζερ, τι πιστεύετε εσείς, ε, είναι σωστή αυτή η δική μου πρόταση, είναι ε, καλός αυτός ο συμβασμός ε, ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες είναι προφανώς η ε, φωνή της σοφίας και θα ήθελα να προσθέσω ένα-δύο πράγματα για να απαντήσω καταρχήν στους συναδέλφους και να σχολιάσω αυτά που είπατε διότι πολλά είπαμε και πολλά επαναλάβαμε γύρω από το τραπέζι. Ναι, μεν ε, ήταν μια τεχνική συμφωνία, εσείς δεν το είπατε κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ, Διατηρήστε και ε, περιφρουρήσατε την, ε, ε, την πολιτική σημασία της συμφωνίας και ότι η Επιτροπή Ίντα ήταν η υπεύθυνη να σταθμίσει εάν ήταν ισοσκελισμένη συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ και αν ήταν επωφελής για την ευρωπαϊκή πλευρά. Στη δεκαετία του 90 δεν θυμάμαι αν ήταν το 96 ή το 97, ο Επίτροπος ΕΣΟ ασχολείται με το θέμα αυτό και υπήρξαν τρία επιπρόσθετα πρωτόκολλα τα οποία περίφθησαν από το Κοινοβούλιο βάσει της εδαφικότητος. Άρα είναι κάτι απολύτως πολιτικό και γι' αυτό και επανελήφθη από την κυρία Ντεσέν. Ε, δεν έχω την ε, παράγραφο δεν έχω την παράγραφο που ανέφερε η Επιτροπή μπροστά μου αλλά εγώ έχω μία νομική γνωμοδότηση η οποία είναι αντίθετη δεν μπορώ λοιπόν να το αφήσω έτσι και όπως είπατε κι εσείς ε, δεν ε, υπάρχει τρομερή βία ξέρω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θέλουν να προχωρήσει αυτή η συμφωνία αλλά αφού δεν έχουμε το μαχαίρι στο λαιμό από πλευράς χρονικής και η ίντα ούτως ή άλλως ε, πρέπει να γνωμοδοτήσει και να αποφασίσει, νομίζω ότι είναι απλή λογική και αυτό δεν είναι μία καθυστέρηση διότι ουσιαστικά θα κινηθούμε σε δύο παράλληλες πορείες η Επιτροπή Ίντα και εμείς. Τώρα, το να συζητήσουμε και να σταθμίσουμε την πολιτική διάσταση με την κυρία Άστον και να ξανασυζητήσουμε το θέμα αν υπάρξει συμφωνία, εγώ το δέχομαι διότι αυτά που είπατε περί πολιτικής συμβιβαστικής λύσης κύριε Πρόεδρε δείχνει ότι είσαστε ένας διαλλακτικός άνθρωπος. <clears throat> Πρέπει όμως αυτό το πρόβλημα να το εξετάσουμε εις βάθος και πολιτικά ε, και νομικά και όχι σαν ένα απλό τεχνικό έγγραφο το οποίο πρέπει να κυρώσουμε διότι είναι αντίθετο στο ότι κάνουμε σε αυτό το τομέα και η Μαρετήλ Γιέκ το παραδέχτηκε ε, είπε ότι, είπε ότι εγώ ονειρευόμουν αλλά δεν ονειρεύω όταν λέω ότι ό,τι ε, συμφωνούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, <clears throat> λαμβάνει υπόψη ότι οι τρεις τομείς πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Οπότε ευχαριστώ τον Πρόεδρο ο οποίος το υπενθύμερεσε και το έλαβε υπόψη όταν παρενέβη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα δηλαδή κάνω την εξής πρόταση. Να κατατεθεί σχέδιο έκθεσης. Βεβαίως ε, θα πρέπει να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για το κατά πόσον θα καταθέσουμε γνωμοδότηση όχι. Αυτό θα το αποφασίσουμε κάποια στιγμή. Μπορούμε αν θέλουμε να έχουμε χρηματοδότηση, μπορεί και όχι. Εγώ θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει, να παρακολουθήσουμε οπωσδήποτε τι ε, πολιτικές ε, διαδικασίες και να δούμε ε, τι γίνεται με την Ίντερ, ε, πώς είναι το δικό σου χρονοδιάγραμμα, κατά πόσον μπορούμε να έχουμε ένα ψήφισμα. Και έτσι λοιπόν Κυρία Ντεκάιζερ, θεωρώ ότι αυτό που έχει νόημα είναι τις επόμενες ημέρες να καταθέσετε την έκθεσή σας. Ε, θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν μπορούσατε ήδη να μας ε, αναφέρετε κάποια στοιχεία του ψοφίσματος έτσι ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε και με την Ίντε να δούμε τι πιστεύουν εκείνοι. Συμφωνείτε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Θέλω λοιπόν να σας προτείνω την ε, έκθεση μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Ε, στην έκθεση του κυρίου Σαλαβράκου, να περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Σαλαβράκου σχετικά με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ε, κυρίως για τη Μεσόγειο. Μάλλον όχι, λέει ο να μην το συζητήσουμε σήμερα αυτό. Ε, να παρακαλέσουμε τον κύριο Σαλαβράκο να μας κάνει μία σύντομη εισήγηση για τρία λεπτά και την επόμενη φορά όταν θα έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες θα έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Συμφωνείτε? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η κυρία Λούνατσεκ. Ναι, αλλά ίσως ε, μπορούμε να προτάξουμε τι ε, ψηφορίε, γιατί ξέρετε έχουν έρθει πάρα πολλοί εδώ για ψηφορίε. Ε, ναι, αλλά είπα στον κύριο Σαλαβράκο, λέει ο πρόεδρος, τρία λεπτά. Δεν είπα να πάρετε όλοι το λόγο στην τοποθέτηση του κύριου Σαλαβράκου. Ε, κοιτάξτε, ο κύριο Σαλαβράκο είχε την καλοσύνη να παρετηθεί από τη συζήτηση. Τον παρακαλέσαμε ε, και το δέχτηκε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να κάνει ήδη τώρα κάποιες παρατηρήσεις, γιατί ήδη μετά από τρεις ημέρες ε, θα υπάρχουν κάποιες εξελίξει. Κύριε Σαλαβράκο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή κατάγομαι από την Ελλάδα, ξέρω και έχω συνηθίσει στις περικοπές. Όπου είναι λογικά τα πράγματα, τα περικόπτουμε από μόνοι μας. Και δεν θέλω να κουράσω τους συναδέλφους. Ε, στην περιοχή της Μεσογείου υπάρχουν πολλές δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ε, με το βέλτιστο τρόπο μέσω μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής ε, και αυτό όπως ξέρετε έχει αποφασιστεί στην συνάντηση της Αγκώνας το 2010 όπου το Συμβούλιο και Κοινωνίου που αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των Χαρών Μελών εξέδωσε δήλωση που υποστηρίζει την πρόταση για την μακροπεριφέρεια. Μέχρι τώρα υπάρχει η στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα σαν μακροπεριφέρεια που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και η μακροπεριφέρεια του Δούναβη. Ε, στο σχέδιο γνωμοδότησής μου, όπως είπα, εξέτασα ειδικά την περιοχή Αδριατικής και Ιωνίου, το έδαφος του οποίου περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία, Ζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία. Αυτές οι χώρες έχουν τη Μεσόγειο θάλασσα ως το σημαντικότερο στοιχείο κοινή κληρονομιάς, περιλαμβάνεται δηλαδή παράκτια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψήφιες ενδυνάμει χώρες η περιοχή εκτός των υδάτων εκτείνεται σε 450.000 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει πληθυσμό 60 εκατομμύρια. Ε, πρώτα απ' όλα για να διευκολύνω την συζήτηση και τους συναδέλφους που θα θέλανε να πάρουν το λόγο και δεν μπορούν λόγω του χρόνου ε, είμαι διαθέσιμος και ανοιχτό σε οποιοδήποτε τροπολογία θα θέλουν στην έκθεσή μου αυτή. Ε, ιδιαίτερα σημεία σημαντικά τα οποία θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να απασχολήσουν τη σκέψη μας είναι το θέμα της υπεραλίευσης και της προστασίας των θαλασσίων πόρων στη Μεσόγειο. Η θάλασσα είναι ένα το σύστημα όπως ξέρετε το οποίο έχει σχεδόν στην περιοχή αυτή μια κλειστή λεκάνη με χαμηλό ποσοστό ανανέωσης του νερού που συνδέεται με το Ιόνιο Πέλαγος και τη Μεσόγειο. Επίσης θεωρώ σημαντική την ανάπτυξη της μακροπεριφερειακής στρατηγικής, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο ενώπιση των γεγονότων που εξελίχθηκαν στις νότιες ακτές της Μεσογείου, που θα πρέπει να αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών ε, πολιτικών γειτονίας η παγκόσμια τρομοκρατία, η παράνομη μετανάστευση, η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, η πειρατεία, η παράνομη αλήψη αποτελούν μερικές από τις κοινέ προκλήσεις των κρατών της Μεσογειακής Λεκάνης. Ήδη έφτασα τα τρία λεπτά κύριε Πρόεδρε και σταματώ εδώ για να αποδείξω ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε να επιτυχάνουμε στις περικοπές. Θα στενοχωρήσω τους συναδέλφους μου βέβαια και τους συνεργάτες μου που έχουν κάνει μια μεγάλη δουλειά, αλλά νομίζω θα ευχαριστήσω όλους εσάς και θα σας πείσω ότι το μελλοντικό μας πρόγραμμα θα επιτύχει. Ευχαριστώ πολύ. Kollege. Das ist hiermit versprochen. Πάρα πολύ ωραία αγαπητέ συνάδελφοι. Την επόμενη φορά θα σας δώσουμε και πάλι το λόγο για να μας η εξωτικά. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 6 στις ε, ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας. Wir stimmen jetzt erst ab über den, die Draft Opinion discharge and respect Ψηφίζουμε για, την, για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, της κυρίας ε, Μίτσου Ιτεμπρόκ, ε, η οποία δεν έχει έρθει ακόμα. Εντάξει, δεν πειράζει, επιταχύνει τη διαδικασία. Πάμε τώρα στην ψηφοφορία. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ της τροπολογία υπαριθμών 1, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, τροπολογία υπαριθμών 2, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 3 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 σε δύο τμήματα. Το 1 αφορά την διαγραφή του sometimes unavoidable. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται το deletion, η διαγραφή. Η υπόλοιπη, για το υπέρ του υπολείπου, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία η 5. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 6 παρακαλώ, σε δύο τμήματα. Πρώτα, όσον αφορά το assistance. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και κατόπιν η εφαρμογή των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Κύριε Ντεκάιζερ, μισό λεπτό σας περιμένουμε. Die Abstimmung ist geschlossen. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίθηκε 45 υπέρ, ε, ένας κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γιαννάκου. Υπάρχουν παρατηρήσει από ό,τι βλέπω όχι. Ε, ξεκινούμε με την ψηφοφορία υπέρ της ε, τροπολογίας 33 παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η, η 9, τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 38 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Η 38 ηλεκτρονικός έλεγχος. Έληξε η ψηφοφορία. 26 ε, υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 41. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13. Υπέρ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 Τροπολογία 20 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 22-23 αποσύρθηκαν. Πάμε στην συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Λάθος. Και αυτή έχει καταπέσει, λέει ο πρόεδρος. Μισό λεπτό. Η 5. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλω να παρακαλέσω του σοσιαλιστές να κάνουν καλύτερη και μεγαλύτερη χρήση του δικαιώματος τους ε, ψηφοφορίας. Δεν ξέρω, εντάξει. 28 κατά αποχές απολύπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία παρακαλώ. Έκλεισε. 38, μισό λεπτό. Τι ψηφίσατε, ναι. 39 λοιπόν, ναι, μία αρνητική ψήφος και 7 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία εισηγήτρια. Πάμε τώρα. Έκθεση Πρέντα ε, για την έκθεση πρόοδου ε, της Ισλανδίας. Η 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, αποδεκτή. 9 και 10. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρώτη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά Νομίζω το δεύτερο ήταν πλειοψηφία, οπότε ηλεκτρονική επαλήθευση ξεκινά για την τροπολογία 16. Έληξε. Απερίφθη με 18 υπέρ και 29 κατά. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι ήταν η ίδια πλειοψηφία με πριν και απορρίφθηκε ξαναελέγχουμε ηλεκτρονικά ξεκινάμε λίγη 22 υπέρ 25 κατά απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 εντρική είναι. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 έχει διεκπαιρεωθεί το 26 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα μέχρι κάντρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 σε δύο τμήματα το πρώτο μέχρι financial system υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Νομίζω περίφθη. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική η ε, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 52 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροπολογία 3 σε 2 τμήματα το πρώτο τμήμα μέχρι historical rights end ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το ποιος είναι υπέρ των ιστορικών δικαιωμάτων, υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ξεκινά. Λίγη. 26 υπέρ, 22 κατά, ε, ε, εγκρίθηκε. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 58 υπέρ κατά αποχές απορρίφθη 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά θα ξαναελέγξουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία και λίγη. 27 υπέρ, 21 κατά. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Λίγοι. 47 υπέρ, ε, μία αρνητική ψήφος. Ελπίζω και σχετικά με την Ισλανδία να έχουμε εξίσου καλά αποτελέσματα και συγχαίρω τον εισηγητή.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 τη Μεσόγειο, Πετροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές ε, ε, ε, αποδεκτή το, η συμβιβαστική πρώτη πρώτα μέχρι το including Christian communities υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το υπόλοιπο από το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΟΚ για την Μεσογειακό Νότο. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε εις ε, την τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά απερίφθη. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το συνολικό σχέδιο γνωμοδότησης. Ξεκινά. Λίγη. Σαράντα υπέρ, δύο κατά, χωρίς καμία από εκεί συγχαίρουμε την εισηγήτρια, κυρία Ρόβολ. Τώρα ερχόμαστε εις τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης εξωτερικής βοηθείας της Επιτροπής από την έδρα της επιφορισμένης για την παράδοση της βοηθείας αντιπροσωπίεσης. Όποιος κατάλαβε περί τίνος πρόκειται μπορεί να ψηφίσει. Ποιος είναι υπέρ της πρώτης τροπολογίας. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έλεγχος ηλεκτρονικός θέλετε. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 3.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 Είχα προηγουμένω υπολογίσει και τον εαυτό μου μαζί. Δεν είχα υπολογίσει μάλλον τον εαυτό μου μαζί. Οπότε τώρα ψηφίζουμε το σύνολο, αλλά έχουμε ακόμη τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, μόνο δύο είχαν καταψηφίσει. Άρα μην ε, το παρακάνουμε. Τώρα βρισκόμαστε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο. Ξεκινά. Λίγη. Σαράντα πέντε υπέρ, τέσσερις κατά. Ευχαριστώ. Συγχαίρω και τον εισηγητή. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε μία σύντομη διακοπή και θα ξεκινήσουμε αμέσως με την ανταλλαγή απόψεων και την ακρόαση του κυρίου James Moran, προσφάτως οριστέντος επικεφαλής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ενώσης στην Αίγυπτο.